αντίρρηση μέχρι την έγκριση των πρακτικών, θεωρούμε ότι εγκρίνονται αυτές οι διορισμοί. Ο, ε, η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς μας προώθησε ένα διευθυντικό από το Κοινοβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 231 παράγραφος 4 και θα πρέπει να γίνει έτοιμα από πολιτική ομάδα ή από τουλάχιστον 40 μέλη για να ψηφιστεί. Τα πρακτικά θα τα βρείτε λοιπόν δημοσιευμένα και σύμφωνα